Σύμφωνα με τον κανονισμό, η έκθεση ισχύει ως εγκριθήσα αν ζητηθεί από έναν αριθμό βουλευτών, αν ε, ζητηθεί η ε, ψηφοφορία από έναν αριθμό βουλευτών. το επόμενο θέμα είναι η έκθεση Βάιντεν Χόλτσερ,